Allora, Καλημέρα σε όλους. Καλώς επιστρέψετε λοιπόν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Έχουμε διάφορες αλλαγές στη μερίσια διάταξη. Φαντάζομαι ότι θα έχετε ενημερωθεί ότι ε, η επίσκεψη από την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Επιστημών, Παιδείας και Πολιτισμού του Ελβετικού Κοινοβουλίου έχει τροποποιηθεί. Οι βουλευτές από την Ελβετία συνάντησαν την πρόεδρο μας ΠΑΚ χθε το απόγευμα, ιδίω για να συζητήσουν την ελβετική συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus Mundus. Επομένως, το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης έχει διαγραφεί. Η εισηγήτρια για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, η κυρία Κώστα, είναι στη Βενετία σήμερα, τυχερή βέβαια. Έτσι λοιπόν το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Πρέπει να σας πω επίσης ότι καθότι δεν υπάρχει κανένα πήγον ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε μπορούμε να αναβάλουμε ακόμα και το σημείο 9, δηλαδή τη συνεδρίαση των συντονιστών στην επόμενη συνεδρίαση, δηλαδή της 17 Σεπτεμβρίου. Τότε θα λάβει χώρα η συνεδρία των συντονιστών. Μετά τις τροποποιήσεις αυτές λοιπόν, σήμερα το πρωί θα έχουμε μια πολύ σύντομη συνεδρίαση. Σας ε, ζητώ λοιπόν να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη όπως τροποποιήθηκε. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων των 17-18 Ιουνίου καθώς και τις 10 και 11 Ιουλίου 2013. Το σχέδιο πρακτικών της 17ης και 18ης Ιουνίου καθώς επίσης και της 10 και 11 Ιουλίου βρίσκονται στο φάκελο με τα υπόλοιπα έγγραφα της συνεδρίασης. Σας προτείνω λοιπόν να εγκριθούν τα πρακτικά αυτά εκτός και αν υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο, επομένως μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης Στο σημείο 3 θα γνωρίζετε βέβαια ότι ε, δυστυχώς ε, φέτος το καλοκαίρι χάσαμε τον ε, συνάδελφο Μπίσκι που απεβίωσε 13 Αυγούστου σε ηλικία 71 ετών. Ήταν μια πολύ σημαντική φυσιογνωμία στη Γερμανία. Ήταν πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος για πάρα πολλά χρόνια και ήταν μέλος του Γερμανικού Κοινοβουλίου και μετά τις εκλογές το 2009 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο ήταν επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΓΚΟΕ κατά το πρώτο τμήμα της τρέχουσας θητείας. Και ήταν επίσης και αντιπρόεδρος και συμμετείχε προφανώς και στη διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμμετείχε επίσης και στην Επιτροπή μας και θα ήθελα να συζητήσω αυτή τη στιγμή να τηρήσουμε ενό λεπτού σιγή με την άδειά σας, αν συμφωνείτε. Ευχαριστώ πολύ. Σα Σας ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω ότι σήμερα δεν έχουμε διερμηνία σε κάποιες γλώσσες βουλγαρικά, κροατικά, εσθονικά, λιθονικά, λετονικά και μαλτέζικα, πορτογαλικά, σλοβενικά και σουηδικά αλλά ακόμα και για τα Ολλανδικά δεν προβλέπεται διερμηνία. Μάλλον μπορείτε όμως να μιλήσετε Ολλανδικά. Απλώς σας έχετε υπόψη σας ότι δεν παρέχετε διερμηνία σε αυτές τις γλώσσες. Τέταρτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ας περάσουμε στις ψηφοφορίες. Η πρώτη ψηφοφορία έχει να κάνει με τις τροπολογίες οι οποίες ε, παρουσιάστηκαν όσον αφορά τον Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες, πολλές συμβαστικές επίσης. Το Συμβούλιο ενέκρινε μια θέση αρκετά αργά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ορισμένε τροπολογίε χρειάστηκε να τροποποιηθούν, να προσαρμοστούν. Δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Λόκεγκαρντ, και να σα υπενθυμίσω κάτι ακόμα. Παρουσιάστηκαν επίση τρει προφορικέ τροπολογίε. Δίνω πάντω το λόγο στον συνάδελφο Λόκεγκαρντ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε επανέλθει από διακοπές τις οποίες αξίζαμε όλοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους γενικούς εισηγητές αυτής της διαπραγμάτευσης που ήταν αρκετά καρποφόρος, όπως θα δείτε στον κατάλογο. Είχαμε πάρα πολλούς συμβιβασμούς και περιλήφθησαν όλοι. Αν συνεχίσουμε την καλή παράδοση που έχουμε σε αυτήν την Επιτροπή, με, θα έχουμε κονσένσους για πάρα πολλά θέματα. Ε, υπάρχουν ε, τρεις τροπολογίες αρκετά αργά, χτες, αλλά θα επανέλθω σε αυτές όταν ε, θα αρχίσουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να παρατείνω την παρέμβασή μου εδώ. Ευχαριστώ. Ε, Μάλιστα. Έχουμε και αρκετό χρόνο βέβαια αυτή τη στιγμή μπροστά μας, που μόνος μπορούμε να προχωρήσουμε ήρεμα, αργά, για να καταφέρουμε όλοι να ψηφίσουμε γνωρίζοντας τι ψηφίζουμε. Χρησιμοποιήστε παρακαλώ πολύ την ηλεκτρονική σας κάρτα, τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία παριθμών 1. Τροπολογία 5702 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5703 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην ε, τροπολογία 57-98 υπέρ κατά αποχές απορριπτεται 5800 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5801 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5751 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε τώρα στην τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε στο σημείο αυτό την προφορική τροπολογία Επί της συμβαστικής 4 είναι η προφορική τροπολογία, παρακαλώ έχετε το λόγο προφορική τροπολογία όσον αφορά τη συμβαστική τροπολογία 4, να προβλέπονται εδώ πέρα 3 εκατομμύρια όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών. Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική σας τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5714. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5715. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5753. Υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην Τροπολογία 5754 δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, καταπίπτει, μάλιστα με συγχωρείτε, καταπίπτει, επομένως περνάμε στη βασική τροπολογία υπαριθμών 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5724 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 57-25. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασική τροπολογία 11. Έχουμε προφορική τροπολογία. Παρακαλώ, κύριε Λόκικα έχετε το... Yes, just the second one, uh, I would... Δεύτερη προφορική ε, τροπολογία στην 11 ε, για τις ε, votiamo il compromesso. Ψηφίζουμε λοιπόν τη συμβαστική υπαριθμών 11 με την προφορική φυτροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57-55 είναι η επόμενη τροπολογία που θα ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57-28 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ πολύ για την 57-28. Άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Νομίζω ότι είχαμε ολοκληρώσει την ψηφοφορία. Λοιπόν, μπορούμε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο όμως το αποτέλεσμα. 13 υπέρ εγκρίνεται. 57-56, εδώ έχουμε μια προφορική τροπολογία και σε αυτό το σημείο. Ναι προφορική τροπολογία για την 5756 6,3 εκατομμύρια για τις πιστώσεις υποχρεώσεων και πληρωμών. Ψηφίσουμε λοιπόν την 5756 όπως τροποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5730 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5731 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5757 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5734 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57-35 έχει αποσυρθεί. 57 λοιπόν υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 57-37 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 57-38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57-58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57-40 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μάλιστα. Συγχαρητήρια κύριε Λόκεγκάρντα και περνάμε τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Δεύτερη ψηφοφορία όσον αφορά την γνωμοδότηση για το ψήφισμα το οποίο θα συνοδεύει την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 10 Ιουλίου είχε παρουσιάσει ο κύριος Λόγκεγκαρτ τη γνωμοδότησή του. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών ήταν 17 Ιουλίου. Έχουν υποβληθεί 9 τροπολογίες και υπάρχουν και κάποιες συμβαστικές. Μπορούμε να περάσουμε ευθύ αμέσω στην ψηφοφορία. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει αντίρρηση.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 Ας περιμένουμε λιγάκι γιατί υπάρχουν κάποιες συσκευές που δεν λειτουργούν από ό,τι φαίνεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται δύο ψήφοι διαφορά. Περνάμε στην τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 9 άρχεται ψηφοφορία. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί πάντως. Πέρας. Όντως, ναι. Σας ζητώ συγγνώμη. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται τροπολογία 9. Τελική τώρα ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται η γνωμοδότησή σας συγχαρητήρια. Α, κάτι ακόμα, σας ζητώ συγγνώμη. Πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός και η τελική ψηφοφορία. Ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για την τελική μας ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν, ομόφωνα σχεδόν. Συγχαρητήρια σε όλους, σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Δεν ξέρω αν ε, θέλετε να γύρετε τώρα κάποιο άλλο θέμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα σημεία πάντα τα οποία πρέπει να θίξουμε. Πρέπει να σας πω ότι ε, η επόμενη συνεδρίαση μας θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου από τις 9 στο 10.30. Σας ευχαριστώ όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, ναι, το